από το Συμβούλιο μια θέση σε πρώτη ανάγνωση για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διαδικασίες Ε, Ο τίτλο θα δημοσιευτεί στα συνοπτικά πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης. Η τρίμηνη προθεσμία που διαθέτει το Κοινοβούλιο για να αποφανθεί αρχίζει από αύριο 16 Απριλίου 2015. Παρακαλώ συνάδελφοι να αποχωρείτε ησύχως διότι ακολουθεί η επόμενη συζήτηση η οποία θα αρχίσει εμέσως.